Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συνεχίσουμε ουσιαστικά την συνεδρίασή μας την χθεσινή. Θα ξεκινήσουμε με τις συζητήσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Πριν δώσω το λόγο στον Φερχόφστατ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ομάδας πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit, θα μου επιτρέψετε πριν το κάνω να πω ορισμένα θέματα τα οποία έχουν σημασία για την Επιτροπή μας. Η εβδομάδα αυτή είναι μια σημαντική εβδομάδα. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συμφωνία, την πρόταση συμφωνίας να σας ενημερώσω όπως το κάνω και σε όλες τις συνεδριάσεις μας ότι ανάμεσα στην προηγούμενη και τη σημερινή συνάντηση υπήρξαν αρκετές συναντήσεις της ομάδας για το Brexit. Υπήρξαν επίσης και πάρα πολλές επαφές τις τελευταίες εβδομάδες σε διμερές επίπεδο. Να σας ενημερώσω ότι κάποιοι συντονιστές μας ήσαν επίσης προσκεκλημένοι στα σεμινάρια γύρω από θέματα τα οποία εντάσσονται στις αρμοδεότητες της Επιτροπής μας, θέματα διακυβέρνησης, θέματα θεσμικά, θέματα κινητικότητας πολιτών και την παρουσία του Προέδρου, του κυρίου Φερχόφστατ, δηλαδή στην οποία και εγώ ανήκω, να παραπονεθώ ότι οι υπηρεσίες της ομάδας αυτής δεν ενημερώνουν ε, τους συντονιστές της Επιτροπής μας για σημαντικά θέματα. Ε, το θέμα της υπηκότητας, της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη είναι κάτι για το οποίο δεν ειδοποιηθήκαμε ότι συζητήθηκε και φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα σχόλια τα οποία θα επιθυμούσαμε. Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αρμοδιότητα και της ΑΦΚΟ κάποια από τα θέματα της υπηκότητας. Εμείς συζητάμε την εφαρμογή της διαδικασίας που αποφασίστηκε από τους συντονιστές. Θα έπρεπε να είχαμε συνεισφέρει κι εμείς οι προηγούμενες εβδομάδες. Δυστυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην συνεχιστεί η λογική αυτή γιατί ο ρόλος της ΑΦΚΟ κρίνω ότι είναι σημαντικός. Είμαστε υπεύθυνοι για τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης, η οποία θα ολοκληρωθεί κανονικά στο τέλος του 18. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια των συντονιστών σήμερα συζητήσαμε ακριβώς και τα θέματα της ΑΦΚΟ που άπτονται του Brexit για τον επόμενο χρόνο. Προγραμματίζουμε τις συναντήσεις που θεωρούμε χρήσιμο ότι πρέπει να υπάρξουν μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία σύμφωνης γνώμης αυτό σημαίνει ότι όλοι μας θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τα προβλήματα αυτά, τα οποία νομίζω ότι οφείλουμε να μας απασχολήσουν. Ασχολούμεθα και με άλλα θέματα, φυσικά όχι μόνο με τον Brexit, αλλά εδώ θα τελειώσω, δεν θα σας κουράσω άλλο. Και θα ήθελα να μας πει ο κύριος Φερχόφστατ πώς εμπλέκεται ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ε, διεργασίες για το Brexit. Για το πρώτο σημείο το οποίο θέσατε, για τα δικαιώματα των πολιτών, φυσικά ένα κομμάτι θα πρέπει να σταλεί και σε εσά και στους συντονιστές της Επιτροπής σας. Όμως το νέο ψήφισμο το οποίο προετοιμάζουμε και θα επανέλθω σε αυτό, δεν υπάρχουν και πάρα πολλά για τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι κάτι που ασχολείται με τις μελλοντικέ σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, είναι θέματα τα οποία συζητάμε και τα οποία θα περιλαμβάνονται στην Συμφωνία για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Πάντως θα ρωτήσω από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να σας ενημερώσουν έτσι ώστε ο πρόεδρός σας και οι συντονιστές σας ή η προεδρος και οι συντονιστές σας να μπορέσουν να ενημερωθούν και να σχολιάσουν. Θα μου επιτρέψετε, Πρόεδρε, να σας παρουσιάσω τις δραστηριότητες της ομάδας της ειδική για τον Brexit του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν ε, τρεις ροές εργασιακού τύπου. Η πρώτη ροή είναι να μεταφέρουμε την έκθεση προόδου του Δεκεμβρίου σε επίσημο κείμενο για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό επίσημα θα ολοκληρωθεί αύριο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα καταθέσει αύριο, θα αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύριο στα ευρωπαϊκά όργανα και ταυτόχρονα επίσης θα την αποστείλει και στην κυβέρνηση της αυτού μεγαλειότητας ένα επίσημο κείμενο το οποίο θα περιλαμβάνει τις προτάσεις για τη Συμφωνία Αποχώρησης. 100 σελίδες ή 150-160 παράγραφοι οι οποίες με επίσημη νομική γλώσσα μεταφέρουν τις αποφάσεις του μηνός Δεκεμβρίου, της εκθέσεως προόδου του μηνός Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η πρώτη ροή, αν θέλετε, ε, προσπάθειας ε, την οποία κάνουμε. Εγώ θα συναντηθώ για αυτό το θέμα και με τον Μισελ Μπαρνιέ σήμερα τα απόγευμα έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η έκθεση προόδου την οποία βρήκαμε σχετικά ικανοποιητική θα μεταφραστεί πλήρως στο επίσημο κείμενο αποχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Θυμίζω Αποχώρησης, είναι και ένα ειδικό πρωτόκολλο ως προσάρτημα για την Ιρλανδία. Για μας φυσικά υπάρχουν δύο σημεία τα οποία έχουν μεγάλη σημασία. Πρώτον, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών θα στραφεί στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το οποίο δεν θα επιθυμούσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχουμε εκφράσει αυτό και στα τρία ψηφίσματα τα οποία έγιναν δεκτά από την Ολομέλεια είναι το θέμα αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγγνώμη, των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών να μας απασχολήσει μετά από την μεταβατική περίοδο γιατί τότε θα καταστεί πραγματικά ένας γραφειοκρατικός εφιάλτης θα καταστεί μια ανεξέλεγκτη διαδικασία που θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες της Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα γίνει επίσης φοβάμαι και κόλαση για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι θα συνεχίσουν να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς λοιπόν οι ανησυχίες μας για τα δικαιώματα των πολιτών δεν είναι μόνο ανησυχία για τους πολίτες της Ένωσης που ζουν στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγγνώμη, αλλά και για τους ε, ε, Βρετανούς που ζουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν παράδειγμα, εφόσον έχουν την δυνατότητα και τα έγγραφα για να εγκαθίστανται σε μία χώρα, αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τις 27 χώρες της Ένωσης και ταυτόχρονα όπως είπα θα πρέπει να προβλεφθεί μια διαδικασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια διαδικασία απλή, μια διαδικασία θα έλεγα ελαφρά, μια δήλωση αν θέλετε, ε, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες, ε, σαν παράδειγμα για λόγους οικογενειακούς, θα δηλώνονται ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες γύρω από αυτό. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εκφράζουν αμφιβολίες και γι' αυτό ακριβώς οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται σε αυτή τη φάση θα προσπαθήσουν να καλύψουν τις ανησυχίες αυτές. Αύριο λοιπόν εμείς θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια του κειμένου το οποίο επαναλαμβάνω θα κυκλοφορήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Μισελ Μπαρνιέ. Θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα περιλαμβάνει και στοιχεία των τριών ψηφισμάτων τα οποία υιοθετήσαμε ότι η διαδικασία δηλαδή για τους πολίτες της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ελαφρά διαδικασία, ότι θα καλύπτονται όλα τους τα δικαιώματα και τα λοιπά. Και δεύτερον, υπάρχει το θέμα του πρωτοκόλου για την Ιρλανδία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα ανεξαρτήτως της καταλήξεως των διαπραγματεύσεων στο μέλλον, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στους κανόνες, της ρυθμίσεις κτλ. ανάμεσα στην Βόρεια Ιρλανδία και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Δεν θα υπάρξουν διακανονιστικές αλλαγές ανάμεσα στην Δημοκρατία και την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι έτσι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εγγυήσει και για την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και για τη Συμφωνία για την Ελευθεροκοινωνία στα σύνορα και νομίζω ότι θα δώσουμε μάχη για την υπόθεση αυτή ε, στα πλαίσια της προτάσεως για το ειδικό πρωτόκολλο το οποίο θα είναι τμήμα της Συμφωνίας Αποχώρησης. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι απαραίτητο βράχη πρόθεσμα και αυτή τη στιγμή η συμφωνία, η πρόταση μάλλον για το επίσημο κείμενο δημοσιευθεί και κυκλοφορήσει αύριο. Πρώτον να κάνουμε μία αξιολόγηση, αυτό το θέλει και η ομάδα χάραξης πολιτικής, το steering group του Κοινοβουλίου και εσείς ως ΑΦΚΟ έτσι ώστε πράγματι τα τρία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να περιλαμβάνονται πλήρως, να το πω αλλιώς, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη στην Συμφωνία Αποχώρησης. Αυτά είναι για τον πρώτο τομέα δραστηριότητας. Ο δεύτερος τομέας είναι το θέμα της λεγόμενης μεταβατικής περίοδου. Θα γνωρίζετε ότι οι Βρετανικές αρχές και η κυρία Μέη έχουν ζητήσει ήδη για μια μεταβατική περίοδο. Εμείς ενθυμίστε ως Κοινοβούλιο ότι εμείς είχαμε αναφερθεί στην ανάγκη στο πρώτο μας ψήφισμα για μια μεταβατική περίοδο και γνωρίζετε επίσης ότι και το Συμβούλιο έχει ε, υιοθετήσει μια εντολή διαπραγμάτευσης για τις ρυθμίσεις για τη μεταβατική περίοδο στις 9 Ιανουαρίου. και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς έχουμε μια ξεκάθαρη αντίληψη για το τι εννοούμε η μεταβατική περίοδος θα πρέπει να είναι περιορισμένη συγκεκριμένου χρόνου. Η πρόταση η αρχική είναι Δεκέμβριος του 2020. Εμείς στο πρώτο μας ψήφισμα ήμασταν κάπως πιο ευέλικτοι. Λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να υπερβεί τα τρία χρόνια. Αυτή ήταν η πρώτη θέση την οποία είχαμε ως Κοινοβούλιο. Πάντως πέραν αυτού και πέραν των χρονικών ορίων, Ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταβατική περίοδο σημαίνει ότι το πλήρε κοινοτικό κεκτημένο θα εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ίδιοι κανόνε οι ίδιες διαδικασίε θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια τη μεταβατική αυτή περίοδου. Το μοναδικό πράγμα το οποίο θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου είναι ότι δεν θα υπάρχει συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων στα ευρωπαϊκά όργανα. δεν θα υπάρχουν εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κοινοβούλιο, στην Επατροπή, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μάλλον κτλ. κτλ. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούμε με τους στόχους αυτούς. Νομίζω ότι προς ε, όφελος και προς το συμφέρον όλων θα πρέπει να υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία για την μεταβατική περίοδο θα πρέπει, ε, έχει μάλλον υπάρξει και μία πρόταση κειμένου από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κυρίου Μπαρνιέ και υπήρξε και μία πρώτη απάντηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επί της προτάσεως του Μπαρνιέ με πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της ε, νομικής ρύθμισης για την μετάβαση, για την μεταβατική περίοδο. Συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν ε, αρκετά θέματα επί των οποίων υπάρχει διαφωνία για τη μεταβατική περίοδο. Ελπίζουμε οι δυσκολίες αυτές να ξεπεραστούν τις επόμενες μέρες Ε, προς όφελος των δικαιωμάτων των πολιτών. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και γενικά και ο διαπραγματευτής της Ένωσης δεν μπορεί να το αποδεχθεί και το επιβεβαιεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι μιλάμε για το κοινοτικό και κεκτημένο στο σύνολό του, όχι μόνο για τα αγαθάκια της υπηρεσίες, αλλά και για τους πολίτες. Δεν θα δεχθούμε εμείς μετά την, μετα... με την αποχώρηση και πριν τη μετάβαση να υπάρξει μια ειδική μεταχείριση, έκτακτη μεταχείριση για τους πολίτες. Και αυτό γιατί αυτοί οι οποίοι θα πάνε στην Αγγλία μετά από την αποχώρηση και πριν την έναρξη της επίσημης περίοδου μετάφασης ε, γνωρίζουν ότι αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρω ότι ένας κοινό άνθρωπος συνειδητοποιεί το τι συμβαίνει, αλλά αυτό το οποίο δεν μπορεί να συμβεί είναι να διαφοροποιήσουμε την κατάσταση, να πούμε ότι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τα αγαθά, τις υπηρεσίες κτλ, αλλά όχι για τους πολίτες. Ένας πολίτης ο οποίος θα φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρηση, αλλά πριν από την μεταβατική περίοδο, δεν μπορεί να ε, αιτηθεί άδεια παραμονής μόνιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώ λοιπόν κάτι τέτοιο εμεί δεν θα μπορούσαμε να το αποδεχθούμε. Είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει επίσης και πάρα πολλά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα διπλό σύστημα χορήγησης θεωρήσεων ε, παραμονής. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε κάποιες διαφωνίες. Ελπίζω να ξεπεραστούν οι διαφωνίες αυτές. Είναι σαφές ότι η μετάβαση σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα εφαρμόζεται πλήρως και θα καλύψει όλους τους τομείς, όχι μόνο τα αγαθά και τις υπηρεσίες, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέλουμε μια πλήρη διακανονιστική αυτονομία της μεταβατικής περίοδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες διαφορετικές δυνατότητες, αλλά είναι σαφές ότι δεν θα υπάρχει συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Και τρίτον, να πούμε ότι για μας το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν είναι κάτι το οποίο έχει ξεκαθαρίσει και είναι στην τελική του φάση. Ε, δεν θα πρέπει να ε, υπάρχουν δυνατότητες για αλλαγές επί των συμφωνιών αυτών. Γιατί αυτό σημαίνει ότι εμείς ως νομοθέτες θα υποστούμε μια κάποια υποβάθμιση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Εμείς θέλουμε εγγυήσει έτσι ώστε ε, φυσικά οι συμφωνίες μπορεί να αλλάζουν αν χρειάζεται, μπορεί να εξυγχρονίζονται, ένα τέταρτο στοιχείο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε στη μεταβατική περίοδο να υπάρχουν νέες μορφές ελέγχου και επίσης ε, υπάρχει και το θέμα των Διεθνών Συμφωνιών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει μία σε εισαγωγικά το λέω τριμεροποίηση των Διεθνών Συμφωνιών δεν θα πρέπει να την χάνει των ωφελημάτων των νέων εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να υπάρχουν άμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την τρίτη χώρα. Δεν θέλουμε εμείς να καταστήσουμε την διαδικασία αυτή τριμερούς φύσεως ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την λεγόμενη τρίτη κάθε φορά χώρα. Αυτές λοιπόν είναι οι ανησυχίες τις οποίες προς στιγμήν εγώ βλέπω μπροστά μου και θα ήθελα να υπογραμμίσω στην Επιτροπή σας εκφράζοντας για μια ακόμη φορά την ελπίδα ότι θα υπάρξει μια σύντομη συμφωνία για την μεταβατική περίοδο. Αυτό είναι προς όφελος όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών γενικά αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο και για όλους όσους επηρεάζονται από το Brexit με τον ένα τρόπο ή άλλο. Οι προθέσεις λοιπόν τις οποίες έχουμε εμείς σαν ομάδα χάραξης πολιτικής είναι να υπάρξει ένα ειδικό κεφάλαιο για την μεταβατική περίοδο και στο νέο ψήφισμα. Αυτό είναι το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να σας θέσω και εδώ έρχομαι στον τρίτο τομέα δραστηριοτήτων, είναι η μελλοντική σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ήγηκε πλέον η ώρα έτσι ώστε και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταθέσει μία πρόταση επεξεργασμένη πλέον για τον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε την εξέλιξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Το ψήφισμα αυτό Κανονικά προβλέπεται με τον εξή τρόπο. Προ στιγμή βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας, σε συνεργασία με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα σας πω πώ ακριβώς το κάνουμε. Δεύτερον, αυτή στιγμή κατατεθεί το ψήφισμα την 7η ή την 8η Μαρτίου στην διάσκεψη των Προέδρων, όπως κάνουμε με κάθε ψήφισμα για το Brexit. Η διάσκεψη των Προέδρων είναι αυτή η οποία αποφασίζει τελικά για την κατάθεση στην Ολομέλεια. Μετά θα πάει στην Ολομέλεια την 13η ή 14η Μαρτίου. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι αν θέλετε στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα που θα πρέπει να υιοθετηθούν στις 23 Μαρτίου. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία Νομίζω ότι είναι χρήσιμο και απαραίτητο να κατατεθεί ένα ψήφισμα, να υιοθετηθεί από την Ολομέλεια, να συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η εκκίνηση, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων, της δεύτερης φάσης των διαπραγματεύσεων, δηλαδή του θέματος των μελλοντικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο οντότητες. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γνωρίζετε ακριβώς πώς έχουμε οργανώσει τα πράγματα. Έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα 10 σεμινάρια Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακριβώς το κάνει και σε συνεργασία με το Συμβούλιο, θα μας δώσει εξηγήσει πώς βλέπει τα θέματα των μελλοντικών σχέσεων σε τομείς όπως το εμπόριο, τις εσωτερικές υποθέσεις, την ασφάλεια, τις μεταφορές, τις αερομεταφορές, την δίκαιη μεταχείριση. Ο κατάλογος εδώ είναι γενικά πάρα πολύ μεγάλος. Έχουμε όλα αυτά τα σεμινάρια που οργανώσαμε με την Κομισιόν και αυτό το οποίο φάνηκε ακριβώς όπως και σε σχέση με το Συμβούλιο το πώς ατενίζουν το μέλλον, ποια είναι τα προβλήματα. Οπότε έχουμε ακόμα ένα σεμινάριο που οφείλει να γίνει, αλλά σε όλα αυτά επίσης έχουν προσκληθεί όλοι οι πρόεδροι των επιτροπών, όλοι οι συναρμόδιες, επίσης οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στη διευθύνουσα ομάδα για το Brexit. το, το άλλο το οποίο κάναμε είναι ότι με την ε, διευθύνουσα στείλαμε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος σε όλες τις ε, μπλεκόμενες επιτροπές. Όπως είπατε, ναι, θα, θα πρέπει να δούμε και με την ΑΦΚΟ, αλλά εκτός το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών, ο, κάθε συγκεκριμένο κομμάτι του σχεδίου του κειμένου το στείλαμε στους πρόεδρους των Επιτροπών και τους είπαμε να συνοηθούν με τους συντονιστές τους και να τοποθετηθούν. Διάφορες προτάσεις και το απόγευμα εκπνέει σχετική προθεσμία. Επομένως, ε, πριν από δέκα μέρες, δεν το στείλαμε χθε έτσι. Δέκα μέρες έχουν περάσει από τότε που το στείλαμε. Ήταν πράσινη εβδομάδα, αλλά δεν υπάρχει πράσινη εβδομάδα για τις διαπραγματεύσεις του Brexit. Ήταν μια φυσιολογική εβδομάδα. Δεν έχει διαφορά. Δεν, έχει, δεν έχουν διαφορετικό χρώμα εβδομάδες στις διαπραγματεύσεις μας. Οπότε, επί τη βάση των όσων μας πούν οι συντονιστές και οι πρόεδροι των επιτροπών, Και δεν μιλούμε τώρα για σχεδόν όλε τι επιτροπέ ότι είναι συναρμόδιε. Επί τη βάση αυτών, επομένω, θα συντάξουμε ένα νέο κείμενο, θα το διαβάσουμε στην διάσκεψη των Προέδρων και 7 ή 8 Μαρτίου θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή στην διάσκεψη των Προέδρων. Η βασική αρχή βασικη τωρα την οποία θέλουμε να προωθήσουμε είναι ότι για τις μέλουσες σχέσεις μας θέλουμε να ισχύσει το άρθρο 8 και το άρθρο 217 της συνθήκης. Και θεωρούμε ότι μπορεί να διαρθρωθεί η συνεργασία σε τέσσερις πυλώνες ε, εμπόριο οικονομία, δεύτερον καινοτομία, θεματικά είτε αερομεταφορές ε, ή άλλου είδους συνεργασία. Θεματική, θεματική. Τρίτος ε, πυλώντας, συνεργασία σε επίπεδο ιστορικής ασφάλειας, αλλά και, και συνεργασία στην εξωτερική πολιτική. Άρθρο 8, το 217. Και αυτά αποτυπώνουμε στο ψήφισμα, τις βασικές αρχές, τις κόκκινες γραμμές, αλλά με θετικό τρόπο. Δεν έχουμε διατύπωση που να αναδεικνύει τις κόκκινες γραμμές και αρνητικότητα. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτή την γενική εικόνα, αποτύπωση του τοπίου, το πώς θα έχουμε αυτή την στενή μέλουσα σχέση με θεμέλιο τις βασικές αξίες της Ένωσης. Αυτά τις αμέσως εβδομάδες και περιμένουμε τώρα την αντίδραση των επιτροπών για τα διάφορα κεφάλαια, τα διάφορα άρθρα του ψηφίσματος. Οπότε είπαμε ότι θα διαβάσουμε το κείμενο στη των Προέδρων 13 και 14 Μαΐου κατά την Ολομέλεια. Έτσι έχουν τα πράγματα τώρα, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Γίλη, κυρία Χιούμνερ και τώρα οι συντονιστές. Πρώτος ο κύριος Σέπφλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Γκί που κάθεται στο πίσω έδρανο που μας ενημέρωσε για το πώς έχουν τα πράγματα και για το προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα. Ε, πρόκειται για το πώς θα δημιουργηθούν οι μέλουσες ε, σχέσεις μας με την Βρετανία. Επ' αυτού θέλω να σας θέσω τα εξής δύο. Έχετε σκεφτεί τα περί επιλύσεως των διαφορών. Είναι σαφές ότι κατά τη μεταβατική περίοδο οι ισχύοντες μηχανισμοί πρόκειται να εφαρμοστούν. Αλλά στο μέλλον. Τι θα γίνει. Οι δύο πλευρές δέχονται να συνεχιστεί αυτή η ρύθμιση. Μας αναφέρατε το άρθρο 8. Βλέπω τώρα εδώ στο κινητό μου τι ορίζει Θα πρέπει να αναπτύξει ειδικέ σχέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ευημερία και καλέ δονικέ σχέσει επί τη βάση των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει, ορίζει το άρθρο Μα ακριβώ το αντίθετο θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλει να απομακρυνθεί από αυτέ τι θεμελιώδεις αξίες. Οπότε προς τα πού πάει το πράγμα. Τι λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει η Πρόεδρος και την την κυρία Μπρέσο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Γκί. για αυτή την τόσο πλήρη αποτύπωση του τοπίου. Γενικώ συμφωνώ ότι πρόκειται για τα στοιχεία αυτά τα οποία πρέπει να υπόψη μας για να οργανωθούμε και επί τη βάση των διαπραγματεύσεων εσείς ξέρετε καλύτερα από ότι εμείς που είμαστε απ' έξω ποια κατεύθυνση θα πάρουν τα πράγματα με τον Βασίλειο γιατί το έργο το οποίο ε, εμείς προσπαθούμε να επιτελέσουμε είναι λίγο στο σκοτάδι. Τι ξέρουμε. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, Καναδά, Ελβετία, αυτά ξέρουμε. Και εργάζομαι στην Επιτροπή των Σχέσεων με την Ελβετία και δεν καταλαβαίνω με τον Καναδά και τον ΕΟΧ, έχουμε στη μέση την Ελβετία. Αυτό είναι ε, ε, λίγο χαοτικό. Οι σχέσεις μας δηλαδή με την Ελβετία είναι λίγο χαοτικές και το κοινωτικό κεκτημένο συνεχώς επικαιροποιείται επί τη βάση των αποφάσεων που λαμβάνουν εκείνοι. Έχουμε συνεχείς ρυθμίσεις σε αυτές τις σχέσεις ε, έχουμε συνεχείς μονομερείς ε, τροποποιήσεις αυτών των σχέσεων οπότε δεν μπορώ να καταλάβω ε, κατά ποιο τρόπο πάμε τώρα για έναν μέσο όρο πάμε δηλαδή ε, να βρούμε τη, τη μέση οδό μεταξύ σχέσεων με Καναδά και σχέσεων με τον ΙΟΧ κάτι που να το καταλάβουμε εμείς είμαστε έξω από το χώρο Και κάποια στιγμή θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να δώσει άργα και ωστά για το τι σκοπεύουν να κάνουν, τι σχέσεις θέλουν για το μέλλον. Για τα οικονομικά βέβαια θα πρέπει να δούμε για τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολα. Αλλά συνεχίζει να εκκρεμεί το θέμα για όλα αυτά για τα οποία θα συνεχίσουμε να έχουμε σχέσεις. Πώς θα εξαιρεθεί το κεκτημένο. Είναι τα προβλήματα. Εκτός αν πάμε για μια απλή εμπορική συμφωνία. Αλλιώς. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ε, έχουμε αυτόματη προσαρμογή στο κεκτημένο για τις σχετικές χώρες. Άρα τι θα γίνει. Αλλά όπως είπαμε είναι λίγο χαοτική η ρύθμιση με την ε, Ελβετία. Άρα θα πρέπει να δρομοποιηθεί και το κοινοτικό δίκαιο για όλα αυτά. Και πώς θα γίνεται αυτό, κάθε φορά θα υπάρχει κάποιο είδου συμβατική ρύθμιση ή θα υπάρχει αυτόματη προσαρμογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η κυρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το θέμα της διαφάνειας και το θέμα της ευελιξίας. Η ευελιξία καταρχήν όσον αφορά την μεταβατική περίοδο. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μία συμφωνία η οποία θα σέβεται και των δύο πλευρών τα συμφέροντα. Αμοιβαίος σεβασμός λοιπόν και φυσικά αυτό που μας παρουσίασε ο κύριος Φερχόφστατ μου φαίνεται λίγο άκαμπτο σαν προσέγγιση. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της μεταβής, μεταβατικής περίοδου θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να σέβεται το κοινοτικό κεκτημένο χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή θα είναι μια χώρα που θα έχει μόνο υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα. Έχω την εντύπωση ότι εν ώψη των μελλοντικών σχέσεων που θέλουμε να δημιουργήσουμε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι προς συμφέρον και των δύο πλευρών να δείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε πιο ανοιχτοί και να δείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Δεύτερο, η διαφάνεια. Δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλει την άποψή του στην Επιτροπή και το Συμβούλιο πριν οι δύο αυτοί θεσμοί, τα δύο αυτά θεσμικά όργανα που είναι αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις να καθορίσουν τη θέση τους. Εάν η Ευρωπαϊκή, αν θέλετε, <clears throat> θέση του Κοινοβουλίου και ο κύριος Φερχόφστατ θέλει να καθορίσει τη δική μας θέση αυτόνομα, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή αυτόνομα, αυτό θα πρέπει να γίνει νωρίς και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να μιλήσει με τη δική του φωνή. Το σχέδιο ψηφίσματος λοιπόν σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι έτοιμο εγκαίρος για να μπορέσουμε και εμείς να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Φαερχόφστατ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση των προοπτικών και την παρουσίαση αυτών που γίνονται στην ομάδα που ασχολείται με το Brexit. Έχω κάποια μηνύματα. Πρώτον, αύριο γίνεται μια μονομερής κίνηση από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αγνοεί πλήρως τις ανακοινώσεις της Πρωθυπουργού της Βρετανίας την Παρασκευή. Σε μια κανονική διαπραγμάτευση, οι δύο πλευρές πορεύονται ταυτόχρονα και ακολουθούν μια κοινή πορεία. Πολλά από τα σημεία που μας αναφέρατε σίγουρα θα απαντηθούν την Παρασκευή, είμαι σίγουρη εγώ ότι θα απαντηθούν, αλλά σήμερα ουσιαστικά εγείρονται τα σημεία αυτά γιατί αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει μονομερώς. Έχω τέσσερις ερωτήσεις. Η πρόθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταπέσει η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη θέση παίρνετε. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά ότι δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακούσατε τις προτάσεις των εργατικών θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει την πίτα και να την φάει ολόκληρη. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν θα δεχόσασταν την άποψη ότι το Βέλγιο είναι μια απικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάτι τέτοιο διαφαίνεται εάν υλοποιήσουμε αυτά που λέτε. Υπάρχουν τέσσερα άτομα τα οποία εκπροσωπούν το Ηνωμένο Βασίλειο. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτό που προτείνουν σήμερα οι εργατικοί είναι ένα ισορροπημένο σενάριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Φερχόφστατ για την περίληψή του. Εγώ θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτό που μας περιγράφεται σαν το πρωτόκολλο που αφορά την Ιρλανδία και την Βόρεια Ιρλανδία. Είπατε ότι για τη Βόρεια Ιρλανδία δεν θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές ρυθμίσεις μεταξύ της Δημοκρατίας Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Παρεμβαίνεται στις εσωτερικές υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Και κάτι που είναι επίσης απαράδεκτο και δεν μπορούμε να το δεχθούμε είναι ακριβώς η θέση που είχατε και θεωρήθηκε απαράδεκτη μεταξύ Ισπανίας και Καταλωνίας γιατί ξαφνικά υιοθετείται άλλη θέση όσον αφορά το θέμα της Ιρλανδίας. Η κυβέρνηση του Δουβλίνου σαφώς και εδώ έχει μία πολύ συγκεκριμένη θέση. Καταλαβαίνετε ότι οι θέσεις που πρεσβεύετε θα είναι καταστροφικές για τη Βόρεια Ιρλανδία. Και ξέρετε ότι οι εξαγωγές της ε, δημοκρατίας της ε, Δημοκρατίας Ιρλανδίας είναι πολύ πιο σημαντικές στο Ηνωμένο Βασίλειο από ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τέτοιου είδους προτάσεις μπορεί να είναι καταστροφικές και για την Δημοκρατία της Ιρλανδίας ακούμε ότι το κείμενο αυτό δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ε, στον τύπο διαρροές πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικών κομματιών αυτού του κειμένου. Μπορείτε να μας πείτε εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει και θα συνεχίσει να έχει τέτοιου είδους ε, θέσεις και εάν η συμφωνία θα μπορέσει κατ' επιλογή και εκεί που συμφέρει μία από τις δύο πλευρές να υλοποιηθεί και αλλού να τροποποιηθεί. Αναφέρομαι στην συμφωνία του Δεκεμβρίου. Άλλη ερώτηση. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο Συμβούλιο του Μαρτίου, τουλάχιστον όσον αφορά αυτά που θέλετε να δημοσιεύσετε αύριο αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, ο Μαξ Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι η συμφωνία μετάβασης θα είναι μια μεικτή συμφωνία. Δηλαδή θα υπάρχει ο κίνδυνος ένα κράτος μέλος, κάποια μέλη, να αποφασίσουν, γιατί έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, να υποβάλουν ε, τις αντιρρήσεις τους και να μην κυρώσουν τη συμφωνία. Άρα δεν θα είναι εγκαίρος έτοιμη αυτή η μεταβατική συμφωνία. Μπορεί να υπάρχει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα προβλήματα λειτουργίας αυτής της μεταβατικής συμφωνίας. Έχετε κάποια άλλη εναλλακτική λύση σε περίπτωση που προκύψουν τέτοιου είδου προβλήματα. Ποιο είναι αυτό το plan B το οποίο έχετε, εάν υπάρχει ένα τέτοιο plan B. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει μία έντονη αντιπαράθεση και ένα μη ομαλό Brexit του χρόνου του Μάρτιο. Θέλω επίσης να αναφερθώ στις προθεσμίες που δώσατε για την μεταβατική αυτή περίοδο. Μπορείτε να μου πείτε κάτι παραπάνω ποια θα είναι η διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου και αν αυτό που προβλέπετε είναι ρεαλιστικό. Θα προλάβετε δηλαδή να διαπραγματευτείτε όλες τις πτυχές αυτής της συμφωνίας θα έχετε αρκετό χρόνο, παραδείγματο χάρη, για να ενημερωθούν και να είναι έτοιμοι όλοι οι υπάλληλοι στα τελωνία, στα, στον ε, τομέα της υγείας, παραδείγματο χάρη. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν σημαντικές πιέσεις για να μειωθεί αυτός ο χρόνος ε, της και η διάρκεια της μεταβατικής περίοδου. Επίσης, όσον αφορά την υλοποίηση της μεταβατικής συμφωνίας, εμείς ε, οι πράσινοι ανησυχούμε γιατί παρόλο που υπάρχουν κάποιες εγγύσει, ότι δηλαδή θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ε, κανόνες και η νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον στη Μεγάλη Βρετανία, ανησυχούμε, διότι αν δεν υπάρξει μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι πραγματικά θα υλοποιούνται όλα αυτά, θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή θα υπάρχουν νόμοι, θα υπάρχει νομοθεσία περιβαλλοντολογική, όμως δεν θα εφαρμόζεται. Το έχετε επεξεργαστεί αυτό το κομμάτι της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας στις διαπραγματεύσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Φερχόφστατ για τις πολύ σαφείς οδηγίες που μας έδωσε για τα επόμενα βήματα. Και εγώ έχω η συμφωνία αποχώρησης και η δήλωσή σας αύριο είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαίρομαι που άκουσα τα σχόλιά σας για το πρωτόκολλο που αφορά την Ιρλανδία και η δέσμευσή σας ε, για την διασυνοριακή αυτή περιοχή. Όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει σήμερα συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Πώς θα προχωρήσουν. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Πρέπει πρώτα να υπάρξει ολοκλήρωση της μεταματικής συμφωνίας και μετά να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για την αποχώρηση. Ή μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα. Όσον αφορά την μελλοντική εταιρική σχέση, σίγουρα θα υπάρξουν ε, πολλές ερμηνείες και γι' αυτό με ενδιαφέρουν οι απαντήσεις σας. Πώς μπορούν, αν θέλετε, να είναι πολύ στενές οι μελλοντικές μας σχέσεις, ενώ θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω να επικρατήσει η γλώσσα και η φωνή της συνένεσης και όχι της αντιπαράθεσης. Τώρα, για τα εσωτερικά μας θέματα. Γνωρίζω ότι ο Μάρτιος, ε, ο Μάρτιος του 2018 είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά ο Μάρτιος του 2019 είναι ακόμα πιο ε, ανησυχητικός. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που να αναλάβετε. Πρόεδρος, επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν ε, να κάνουν ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ να είστε σύντομοι. Κύριος Φόξ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φερχόστατ που μας ενημερώσατε. Και εγώ έχω τρεις ερωτήσεις και θα ήθελα να σας τις κάνω. Πρώτον, τα δικαιώματα ψήφου στις τοπικές εκλογές των Βρετανών και μη Βρετανών κατοίκων της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Ευρωπαίοι που διαμένουν στην ε, Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να διατηρήσουν τα δικαιώματα ψήφου στις τοπικές εκλογές, αλλά θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαιότητα. Ποια είναι η στάση, γιατί εδώ φαίνομαι ότι διαφέρει η στάση του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, τα δικαιώματα των σύζυγων Βρετανίδων που έχουν δηλαδή παντρευτεί με πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης των Βρετανών, παραδείγματος χάρη, σκέφτομαι ένα παράδειγμα, που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι παντρεμένοι με, παραδείγματος χάρη, Βελγίδες. Εάν αυτό το ζευγάρι θέλει να φύγει, παραδείγματο χάρη από τη Μεγάλη Βρετανία και να ζήσει κάπου, να εγκατασταθεί κάπου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίθετο, το ζευγάρι το οποίο θέλει να φύγει από το Βέλγιο και να ζήσει στην Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει πιστεύω να υπάρξει μια συμφωνία που να αφορά τις συζύγους και την οικογένεια ε, αυτών των ε, Ευρωπαίων και Βρετανών πολιτών. Και μια άλλη ερώτηση που έγινε από την Time Dodge. Μιλήσατε για την ε, δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βρετανική κυβέρνηση σαφώς και έχει δεσμευτεί να σεβαστεί τη συμφωνία του Μπέλφαστ. Αυτό όμως που εσείς λέτε είναι καθαρά κάτι που μας απομακρύνει από την πραγματικότητα. Από την ημέρα που θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξουν όλες αυτές οι ρυθμίσεις. Και βεβαίως μιλήσατε για την δέσμευση να μην υπάρξουν σκληρά σύνορα, όπως τα λέμε. Μπορείτε να μας πείτε ε, πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Θεωρώ ότι οι θέσεις σας είναι καθαρά μη ρεαλιστικές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ για όλα όσα μας είπατε. Έχω δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Η μία είναι, είπατε ότι δεν θα υπάρξει ειδικό καθεστώς για τους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, αυτούς που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εννοείται ότι τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φτάσουν μέχρι την τελευταία μέρα της μεταβατικής περίοδου θα είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά των υπολείπων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό όσον αφορά την καταχώρησή τους ε, σε Μητρώα κτλ. Όλες δηλαδή οι διαδικασίες που τους υποχρεώνει το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουν θα είναι οι ίδιες με αυτές των ήδη εγκατεστημένων πολιτών. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου βεβαίως δεν θα υπάρξει θεσμική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο αυτό θα ισχύει αυτόματα κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Μπροκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον Κίφερ Χόφστατ. Εγώ συμφωνώ πολύ με την ανάλυση του και έχω κάποιες παρατηρήσεις συμπληρωματικές και κάποιες ερωτήσεις. Ήμασταν μαζί στο Λονδίνο και μιλήσαμε με εκπροσώπους της ε, κυβέρνησης. Το θέμα της ε, Ιρλανδίας. Σαφώς και η συμφωνία του Δεκεμβρίου θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλες αυτές τις πτυχές. Και όπως είπε ο κ. Φόξ, είναι δύσκολο το θέμα αυτό. Εννοείται ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές αυτών που ισχύουν. Δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης ε, συμμόρφωση. Αυτό όμως θα είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια τρίτη χώρα, όπου τα πρότυπα και τα ισχύοντα θα αποκλίνουν μέχρι τώρα, όποτε συνάπτουμε μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και μιας τρίτης χώρας, η ιδέα ήταν τα πρότυπα και η πραγματικότητα σιγά σιγά να συγκλίνουν. Για πρώτη φορά θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα πρότυπα θα αποκλίνουν, θα διαφοροποιούνται και αυτό θα γίνει αν θέλετε με την Ιρλανδία και νομίζω ότι εδώ πρέπει να δείξουμε φαντασία δημιουργικότητα και η συζήτηση, αν θέλετε, που είχαμε με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων, αν θέλετε, έλαβε υπόψη ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε μια συμφωνία για αποχώρηση και όχι για ε, σύνδεση. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφώς και έχει το δικαίωμα να <laughs> υποβάλει τις προτάσεις του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι δικαίωμά μας, δεν είναι κάτι που κάνουμε και μπορεί να ληφθεί υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς και <coughs> μέχρι την Παρασκευή που θα κάνει τις δηλώσεις της η κυβέρνηση. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε τις προτάσεις μας πριν την Παρασκευή. Γιατί να περιμένουμε δύο μέρες μέχρι να αποφασίσει η Βρετανική κυβέρνηση να κάνει τις ανακοινώσεις της. Πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές καλούνται και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που έχει δοθεί να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις προτάσεις της για την αποχώρηση. Και η Βρετανική κυβέρνηση θα κάνει τις δικές της. Νομίζω ότι δεν ε, υπάρχει εδώ σημαντική δυσκολία. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί τόσο πολύ αντιδράτε. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Ελπίζω πραγματικά ότι την Παρασκευή θα βγουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις από αυτές τις δηλώσεις της Βρετανικής κυβέρνησης. Και το θέμα της αντιμετώπισης των διαφορών, της διαχείρισης των διαφορών. Και να αρχίσει πραγματικά η διαπραγμάτευση επί της ουσίας. Το θέμα της μεταβατικής συμφωνίας το θέμα της μεικτής συμφωνίας εμένα δεν με ανησυχεί. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βρει τρόπο να προχωρήσει αυτή η ας πούμε διετής μεταβατική περίοδος. Μιλάμε για 21 μήνες. Εμείς είχαμε προτείνει τρία χρόνια. Αυτή ήταν η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είναι σαφής η συμφωνία όσον αφορά παραδείγματος τα εμπορικά θέματα και να λάβει σοβαρά υπόψη της η Μεγάλη Βρετανία αυτές τις δεσμεύσεις. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μας απασχολεί σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και εδώ δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία, αν θέλετε, τύπου Ελβετίας ή Νορβηγίας. Πρόκειται για δύο χώρες με πολύ συγκεκριμένες θέσεις επ' αυτού. Τελωνιακή Ένωση, εσωτερική αγορά. Αναφερόμαστε σε πολύ συγκεκριμένες συμφωνίες, των οποίων το επίπεδο είναι, αν θέλετε, καλύπτει συγκεκριμένους τομείς και δεν είναι δυνατόν, αν θέλετε, να διαταράξουμε τομείς οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μέχρι τώρα λειτουργούν καλά υπό την προϋπόθεση ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε τη συμφωνία επιλεκτικά. Αυτό δεν γίνεται. Σε συνέχεια τον όσο μας εξήγησε ο κύριος Μπρόκ, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έναν προσανατολισμό προς τα που θέλουμε να πάμε αυτή η συμφωνία. Πέρα από τις εσωτερικές εντάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου των οποίο γινόμαστε μάρτυρες, πέρα από αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λύση θέλει να δώσει στο θέμα. Θα πρέπει να είναι εθνικά κυρίαρχη σχετική απόφαση. Άρα, πρώτη μου συμβουλή, κύριε Φερχόφστατ, είναι η εξή. Θα πρέπει να δούμε τι επιθυμούμε για τις μέλους σχέσεις. Ήδη το Βασίλειο έλαβε μια απόφαση να αποφύγουμε τον πειρασμό να εκμεταλλευτούμε τις εσωτερικές αντιφάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το πώς θα ανακληθεί η απόφαση που έλαβε ο Βρετανικός λαός. Δεν είναι λογικό αυτό. Όμως νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φερθεί με μεγάλη σοβαρότητα στην αναζήτηση επίτευξης συμφωνίας να δούμε πώς θα καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή συμφωνία, για πολλούς λόγους. Εμπορικά, οικονομικά, από πλευρά ασφάλεια, Άμυνα, γεωπολιτική επιρροή, θα πρέπει το Ηνωμένο να μην συμπήξει άλλη συμμαχία υπερατλαντική, το οποίο θα είναι κατά των συμφερόντων μας Μα συμφέρει να έχουμε αγαστέ σχέσει με τη χώρα, επομένω θα πρέπει να επεξεργαστούμε αυτή την ε, πρόταση, την πρόταση του κ. Κόρμπη για το πώ θα επιληθούν οι προστριβές και να είναι μια αξιόλογη συμφωνία και να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα κάνουν και οι Βρετανοί. Είναι θέμα ιστορική πολιτικής, αλλά εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε μια καλή συμφωνία για το μέλλον. Άρα προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Πολύ σημαντικό. Για την Ευρώπη, για το μέλλον. Είναι πολύ κακό να αφήσουμε να προσεγγίσει το Εμένο Βασίλειο της ε, είπα και να αρχίσει ένας ανταγωνισμός σε κάθε επίπεδο οικονομικό. Άρα αυτό θα πρέπει να δούμε, να αναζητήσουμε την καλή συμφωνία. Εμείς αυτό έχουμε προτείνει, το να υπάρχει μια καλή συνύπαρξη στο μέλλον. Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γκίφερ Χόφστατ για τις ενημέρωση που μας έκανε και έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Αυτό που μόλις είπε ο Ραμόν είναι σημαντικό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για την ε, μελλοντική μας συμφωνία θα πρέπει να διαπιστώσουμε εκ των προτέρων και το ξέρουμε ότι θα είναι μια sui generis συμφωνία. Άρα θα πρέπει να εντοπίσουμε εμείς ποια είναι τα κεντρικά σημεία, ποια είναι τα σημεία αυτά που θα πρέπει να λυθούν με έναν ε, επικοδομητικό τρόπο, με έναν τρόπο που να σέβεται ε, κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα. Και θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και διαφάνεια γύρω από αυτές τις κεντρικές, αν θέλετε, ιδέες που είναι σημαντικές για μας και να καταλάβουν οι πολίτες της Ευρώπης γιατί διαπραγματευόμαστε και πού πάμε. Το θέμα της ε, Ιρλανδίας βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να μπούμε σε μία μαραθώνια διαπραγμάτευση και να χαθούμε γιατί εκεί θα χαθεί η διαφάνεια θα πρέπει να επικρατήσει σαφήνεια και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο σε κάθε περίπτωση το νωρίτερο δυνατόν θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ως προς τη μελλοντική αυτή συμφωνία που τελικά θα επικρατήσει. Βεβαίως και μπορούμε να μακρηγορούμε και να συζητάμε επάπειρον, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να υποβάλουμε εμείς με σαφήνεια τις θέσεις μας και αν η Βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να μην είναι σαφής, να καθυστερεί, να αναβάλει, να ε, ζει δηλαδή σε μια αβεβαιότητα, μια αβεβαιότητα η οποία καταστρέφει την αξιοπιστία και τη δική μας και τη δική τους αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών, Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα είναι πραγματικά αρνητικό για όλους μας. Ελπίζω αυτή τη βδομάδα να κάνουμε βήματα προς τη σαφήνεια, προς την δημιουργία ενός κλίματος ε, εμπιστοσύνης, αλλά εμείς η δικιά μας, αν θέλετε, ε, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να εκφράσουμε με ξεκάθαρο τρόπο αυτά που για μας είναι σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ, Γκί. Έχεις το λόγο. Uh, να ευχαριστήσω τον Έλμαρ για τα σχόλιά του. Ήδη έχει δώσει απαντήσεις σε κάποια από τα σημεία τα οποία έθεσαν οι συνάδελφοι. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω λοιπόν. αλλά να ξεκινήσω με αυτά που είπε ο Σόλτς και άλλοι. αυτό είναι και ο στόχος του νέου ψηφίσματος. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει επιτέλους την άποψή του. Όχι να λέμε θα περιμένουμε, θα περιμένουμε και θα περιμένουμε. Να περιμένουμε τι. Θέλουμε μια στενή σχέση ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες θέτει το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούμε να δώσουμε εγγύησει για τις τέσσερις ελευθερίες, εμείς ιδιαίτερα για την ελεύθερη διακίνηση και δεν θα πρέπει να μην λάβουμε υπόψη μας τις κόκκινες γραμμές αυτές. Καιρός θα είναι να ε, εκφραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να δούμε ακριβώς τι θέλουμε, με ποια ε, βάση στη συνθήκη θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την σχέση να δούμε με τα κομμάτια της διαπραγμάτευσης τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε και να πούμε ότι ας δούμε πρώτα πόσο θα περάσουμε στην επισημοποίηση της συμφωνίας αποχώρησης για να αντιδράσουμε. Όχι. Νομίζω ότι τον Οκτέβριο-Νοέμβριο θα πρέπει η διαδικασία αποχώρησης να ολοκληρωθεί και θα έρθει για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα παράρτημα ή χωρίς παράρτημα, εν πάση περιπτώσει θα δούμε ακριβώς, πάντως θα υπάρξει μια πολιτική δήλωση για τις μελλοντικέ σχέσεις. Και επί των μελλοντικών σχέσεων έχουμε κάθε συμφέρον εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωρίζουμε λεπτομέρειες έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ακριβώς τον μέλλον των σχέσεων αυτών. Δεν μπορούμε απλά να γενικολογούμε. Αυτός είναι και ο λόγος λοιπόν για τον οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο τις επόμενες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει θέσεις για το θέμα των μελλοντικών σχέσεων και όχι μέσα σε μία ή δύο παραγράφους, αλλά να εκφράσουμε σε επίπεδο λεπτομέρειας το πώς βλέπουμε τη συνεργασία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ένωση. Ως προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει και η πρόβλεψη ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Μιλάμε για μια εταιρική σχέση αλλά με διαφορετικές συμφωνίες και διαφορετικά κεφάλαια. Θα υπάρξει προφανώς μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα πρέπει να υπάρξει επίσης ε, και ε, συμφωνία για θεματολογικές συμφωνίες με διαφορετικές ρυθμίσεις, σαν παράδειγμα το ΕΡΑΤΟΜ. Για την ΕΡΑΤΟΜ δεν μπορούμε να κάνουμε την ίδια ρύθμιση που θα κάνουμε για το Εράσμους ή για το Horizon 2020, θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές ρυθμίσεις, το ίδιο και για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής ασφάλειας κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια σειρά συμφωνιών που θα ξεκαθαρίζει σύμφωνα με το άρθρο 8 και το 2.17 τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να τα εντάξουμε αυτά σε ένα λογικό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι εφαρμόσιμο το άρθρο 8 δεν νομίζω ότι η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει από τις αξίες της Ένωσης, θα αποχωρήσει από την Ένωση. Εγώ είμαι παλιοχαρακτήρας, θα μπορούσα να τα συγκρίνω αυτά με το τι γίνονται στην Πολωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το κάνω. Αυτό ήταν αστείο, μη με παρεξηγείτε. Αλλά ήταν αστείο βέβαια, το οποίο κρύβει ίσως εν μέρη μια πραγματικότητα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να αλλάξουμε τις αξίες της Ένωσης, αφήνει τους δομές της Ένωσης, αφήνει την Ένωση η Μεγάλη Βρετανία, όχι τις αξίες όμως της Ένωσης. Τώρα για τις μελλοντικές σχέσεις και αυτά τα οποία είπε η Μεσέντες. Εγώ αναφέρθηκα ήδη στις κόκκινες γραμμές που καθιστούν ε, την ολοκλήρωση κάποιων μέτρων για την εσωτερική αγορά ανέφικτη κτλ. Από πλευρά των Βρετανών, ο κύριος Τάσκ το έχει πει αυτό, εγώ επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε, είναι ψευδέστηση να πιστεύει κανείς ότι θα λυθούν τα προβλήματα με την φιλόδοξη διαχείριση της διαφορετικότητας. Ε, τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει, είναι κάποιες λέξεις βέβαια, οι οποίες προσπαθούν να καθορίσουν τα λεγόμενα τρία καλάθια που θέλουν οι Βρετανοί. Το πρώτο καλάθι με τομείς πολιτικής τους οποίους υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεύτερο καλάθι με διαφορετικές απόψεις για συγκεκριμένες πολιτικές και ένα ενδιάμεσο καλάθι στο οποίο θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο για μια μελλοντική ευθυγράμμιση. Για μας ο τρόπος αυτός με τον οποίο τίθενται τα πράγματα δεν ε, είναι αποδεκτός. Αυτό είναι το λεγόμενο ε, «εγώ αποφασίζω, εγώ διαλέγω» στο πρώτο καλάθι βάζω αυτά που με βολεύουν, στο δεύτερο καλάθι αυτά που δεν με βολεύουν και στο τρίτο καλάθι βάζω όλα τα υπόλοιπα για τα οποία δεν ξέρω τι θα γίνει. Συνεπώς λοιπόν δεν είναι τρόπος αυτός για να συνεχίζουμε και γι' αυτό όπως είπε ο Τάσκ είναι ψευδέστηση το να πιστεύει κανείς ότι μπορούμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και ελπίζω ως εκ τούτου ότι η κυρία Μέη θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις και θα επιδείξει ότι και από πλευράς ε, Βρετανικής υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις για τις μελλοντικές σχέσεις και ότι είναι απαραίτητο για τη δεύτερη φάση να επιταχυνθούν επιτέλους οι διαπραγματεύσεις. Τώρα, ο Τάσκα αναφέρθηκε επίσης ε, και για τις ε, διαπραγματεύσεις, επαναλαμβάνω, αλλά και τις ε, ε, επόμενες πολιτικές οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Η Μεγάλη Βρετανία θα συνεχίσει να είναι στο Horizon 2020, στο Erasmus κτλ. Ε, δεν σημαίνει μόνο υποχρεώσεις το νέο κεκτημένο. Το ξέρετε και στην Πολωνία αυτή ότι το νέο κεκτημένο δεν σημαίνει μόνο κεκτημένες υποχρεώσεις, αλλά και ωφέλη. Αυτό το οποίο λοιπόν προσπαθούμε να δείξουμε είναι ότι το νέο κεκτημένο μεν θα συνεχιστεί ιδιαίτερα στους τομείς πάνω στους οποίους θα πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις με το Συμβούλιο, με το Δικαστήριο, με την Επιτροπή κτλ. Δεν μιλάμε μόνο για υποχρεώσεις. Το κεκτημένο είναι και πλέον εκτίματα. Το κεκτημένο είναι και ωφέλη. Και τώρα για την Βόρεια Ιρλανδία. Εδώ υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις γύρω από αυτό. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο δεν θέλει να υπάρξουν σκληρά σύνορα, δεν θέλει να υπάρξει μια σκλήρινση των ελέγχων στα σύνορα, Κάποιοι μας κατηγορούν λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει αναφορά στη Συμφωνία Αποχώρησης για την παράγραφο 15 της έκθεσης πρόοδου. Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι επισημοποιούν την Συμφωνία Αποχώρησης λέγουν ότι η παράγραφος 50 αναφέρεται στην αποφυγή ενός εσωτερικού συνόρου ανάμεσα στις δύο χώρες περιοχές και βλέπουν το θέμα αυτό σαν βρετανικό θέμα και όχι θέμα αποχώρησης και συμφωνίας αποχώρησης. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική αυτών οι οποίοι συγγράφουν την συμφωνία αποχώρησης. Η συμφωνία αποχώρησης αναφέρεται σε θέματα αποχώρησης, όχι σε στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες εντάσσονται στις εσωτερικές υποθέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. να πω ότι η μετάβαση θα είναι τμήμα της συμφωνίας αποχώρησης. Δεν θα υπάρξουν δύο διαφορετικά θέματα. Η συμφωνία αποχώρησης θα έχει ένα κεφάλαιο επίσης για την μεταβατική περίοδο. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε από κοινού και εμείς θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσουμε. Τώρα το τι θα συμβεί αν δεν υπάρχει συμφωνία αποχώρησης. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο ε, δεν το επιθυμούμε, δεν θέλουμε να συμβεί, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Ε, φυσικά και θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Αν όχι το Δεκέμβριο του 2020, ε, λίγους μήνες μετά δεν είναι πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ε, η μεγάλη, πολύ μεγάλη περίοδος η μεταβατική και ακριβώς το άρθρο 50 είναι αυτό το οποίο καθορίζει το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούμε. Το ότι η μετάβαση είναι κάτι το εφικτό πάνω στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε. Φυσικά μπορούμε να δούμε και άλλα επιχείρηματα τα οποία υπάρχουν. Όταν μια χώρα εντάσσεται με βάση το άρθρο 49 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί προβλέπονται μεταβατικές περίοδοι. Έχουν, ε, Έχουν υπάρξει επταετής περίοδοι μεταβατικοί. Σαν παράδειγμα το, το κεκτημένο Σέγγεν κάποιες χώρες εξακολουθούν να είναι σε διαδικασία μετάβασης μετά από χρόνια ιδιότητας μέλους. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο να δημιουργεί ένα, μια μονιμότητα θα έλεγα και μια στασιμότητα. Νομίζω ότι μέχρι τρία χρόνια είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να δεχθούμε. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις του κ. Μπαρνιέ, ο οποίος προβλέπει το Δεκέμβριο του 2020 ως προθεσμία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω ήδη απαντήσει στις παρατηρήσεις της κυρίας Μαγκίνης δεν μιλάμε από τώρα μέχρι τον Μάρτιο, αλλά από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Έξι μήνες, μέσα σε έξι μήνες θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την μεταβατική περίοδο, ε, τη συμφωνία αποχώρησης κτλ. κτλ. Ο κύριος Φόξ έχει δίκιο για τα δικαιώματα ψήφου, αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη Ίσως είναι καλή ιδέα το ότι θέλετε εσείς σαν συντηρητικό κόμμα να καθορίσετε τα θέματα της ψηφοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ είμαι φεντεραλιστής, δεν είμαι κατά της πρότασης αυτής, αλλά θα εξαρτηθεί από το τι θέλουν τα κράτη-μέλη. Πάντως είμαστε υπέρ. Έλαβα υπόψη επίσης τις ανησυχίες σας για τους τις συζύγους είναι κάτι το οποίο θα ζητήσω να συζητήσουμε σε σχέση με την ΑΦΚΟ. Για την κυρία Περέρα αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τη λειτουργία του νέου συστήματος Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να δεχθούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζει ένα νέο σύστημα, ε, να ετοιμάσει ένα νέο σύστημα κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου της μεταβατικής. Δεν είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση πρόοδου. Καλύπτεται λοιπόν το θέμα του καθεστώτος των Ευρωπαίων πολιτών που θα ζουν στο μέλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτι το οποίο δεν θα αναφέρεται στα θέματα τα οποία θα περιλαμβάνει η έκθεση προόδου. Αναφέρεστε ας πούμε στη μεταβατική περίοδο και την ονομάζεται εφαρμοστική περίοδο. Αυτό το βρίσκω παράλογο. Τώρα αν χρειάζεται για πολιτικούς λόγους να το κάνετε αυτό και να μιλάτε για implementation period, για περίοδο εφαρμογής, γιατί όχι, αλλά πάντως δεν έχει λογική αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουμε με σωστό τρόπο το νέο σύστημα, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνει είναι ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να πρέπει να υφίστανται ε, διαφορετικά δικαιώματα, μάλλον διαφορετικές ρυθμίσεις για τα δικαιώματά τους από ό,τι σε άλλες, ε, ε, από ό,τι άλλοι πολίτες. Κάποιος ο οποίος έρχεται μετά την αποχώρηση αλλά πριν τη μετάβαση είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχει τα δικαιώματα που θα είχε και πριν από τις αλλαγές και τα ίδια δικαιώματα τα οποία θα έχουν ε, ε, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεγάλη Βρετανία στα πλαίσια του λεγόμενου νέου καθεστώτος. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες ε, πολιτών. Αυτοί οι οποίοι ε, είχαν πάει πριν από την αποχώρηση να έχουν διαφορετικές δυνατότητες με αυτούς οι οποίοι θα πάνε αμέσως μετά την αποχώρηση, να έχουν οι καινούργοι λιγότερες δυνατότητες από τους παλιούς. Όχι, εγώ νομίζω ότι ε, το κεκτημένο είναι κεκτημένο και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε να υπάρχουν εν πάση περιπτώσει διαφοροποίησεις Νομίζω ότι αυτό θα διευκρινιστεί από πλευρά της κυρίας Μέη την ε, Παρασκευή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ανεμπόδαστα την επόμενη ε, είπατε κάτι για το Βέλγιο ως απικία. Και κοιτάξτε, εμάς μας έχουν καταλάβει οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί πρόσφατα και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που δεν μας έχει κατακτήσει κανείς. Ένας από τους λόγους είναι ότι είμαστε μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πριν ε, πραγματικά ε, είχαμε υποστεί την κατοχή πολλών άλλων χωρών. Τελείωσα και Σόφλιν, μην ανησυχείτε. Ο Πρόεδρος. Ε, εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Φερχόφσταθ. Και μάλιστα μου άρεσαν αυτό το οποίο είπατε για την Ουγγαρία. Πάρα πολύ πλήρης η παρουσίασή σας για το πώς έχουν τα πράγματα και τώρα προχωρούμε. Ε, προσωρινά, τελείως προσωρινά έχω αντικαταστήσει την πρόεδρο και να σας κάνω και κάποιες ε, ανακοινώσεις σε λίγο μόλις ε, έχετε φύγει όσοι από εσάς το επιθυμείτε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 Ο πρόεδρο. Νομίζω ότι οποίο ήθελε έχει αποχωρήσει. Οπότε ας συνεχίσουμε. Μετσέντε, αν θέλει. ησυχία. Ανακοινώσεις του πρώτου. Σας διαβάζω το κείμενο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για λόγους τακτικής οι προθεσμοί για τις τροπολογίες όσον αφορά το σχέδιο αγνομοδότησης Ουζεντόφσκι για την νομοθεσία 2016 ήταν για τις 2 Μαρτίου και τώρα παρατείνεται αυτή η προθεσμία και πάει στις 6 Μαρτίου. Α, το άλλο αφορά εμένα, δεν μπορούσα να είμαι εδώ για ιατρικούς λόγους και στη συνέχεια έχουμε το, το μεγαλύτερο Μποτιλιάς με ιστορία των ε, Βρυξελών και γι' αυτό και ε, πρόκειται περί της αναβολής του δικού μου κειμένου όσον αφορά την πρωτοβουλία των πολιτών και να το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Και τώρα συνεχίζουμε. Ο ρόλος των ε, πολιτών ο κύριος ε, Ζντόφσκι είναι ο συντάκτης και συμφώνω με το άρθρο 54 έχουμε συνομιλήσει με την Περιφερειακή Επιτροπή, Ζεσδόφσκι, αλλά και ο κύριος Όλμπριχτ ε, τα έχουν αναλάβει για μας και για την Ρέτζη και είναι σε στενή επαφή την αρχή της διαδικασίας και το σχέδιο του κειμένου υποβλήθηκε προς ε, μετάφραση, είχαμε διάφορα τεχνικά ζητήματα ε, όσον αφορά την ε, διόρθωση διάφορα κείμενα, κείμενα και οπότε έχουμε κάποια κείμενα γαλλικά, γερμανικά, πολωνικά, ουγγρικά. Τα υπόλοιπες μεταφράσεις θα υπάρχουν από την 1η Μαρτίου και ε, έχουν διανεμηθεί κείμενα στα αγγλικά σε όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν διαβιβαστεί στις 20 Φεβρουαρίου από τη γραμματεία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ιζα Ζντόφσκι. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, έχω την τιμή να σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο κειμένου που αφορά τον ρόλο των πόλεων στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα όλους με τους οποίους είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις για να ετοιμάσω το κείμενό μου πρώτα πρώτα τον κύριο Γιάνν Όλμπριχτ ο οποίος έχει αναλάβει την ε, έκθεση από πλευράς της Περιφερειακής Επιτροπής. Και έτσι θα μας βοηθήσει και αυτή η Επιτροπή. Ναι, επίσης, ευχαριστώ και τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες της Επιτροπής μας. Όλους σας ευχαριστώ. για την άτυπη ανταλλαγή απόψεων και για τις παρατηρήσεις σας. Όσα, ε, όσα, είπατε, τέλο πάντων στο βαθμό του δυνατού, τα έχω ενσωματώσει στο κείμενό μου. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτό το θέμα είναι το εξή. Η αναβάθμιση του ρόλου των πόλεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μοναδικός τους ξεχωριστός χαρακτήρας. Γι' αυτά θα σας μιλήσω. Πρώτα πρώτα, η αναβάθμιση του ρόλου τους. Πρώτα πρώτα όλοι οι Ευρωπαίοι παράγοντες έχουν διαπιστώσει ότι για τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών και συμφωνή του είναι κάτι που έχει σχέση με τις πόλεις, οικολογία, μεταφορά, κοινοφιλείς υπηρεσίες, ε, ασφάλεια, καταπολέμηση της ε, περιθωριοποίησης, μετανάστευση, Πολλές φορές η πόλη είναι στο επίκεντρο αυτών των ε, πολιτικών. Άρα θα πρέπει εκεί να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας. Και η νομοθεσία σήμερα θα πρέπει επίσης να σχετίζεται περισσότερο με τις βίλες και με την ε, χωροταξική πολιτική. Άρα, ο πρώτος λόγος είναι αυτός, αυτή η λειτουργία των πόλεων. Δεύτερος ε, λόγος για τον οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα αναβαθμίσουμε περισσότερο τις πόλεις είναι το ότι οι πόλεις έχουν μοναδικές ξεχωριστές δυνατότητες όσον αφορά τον κοινωνικό βίο. Είναι ο χώρος, είναι το, ο τόπος που έχουμε τα μέσα ενημέρωση τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχει δίκτυο πόλεων με τέτοιες ε, ιδιότητες. Επομένως, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά των πόλεων για τη λειτουργία της Ένωσης. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου προβαίνω σε κάποιες προτάσεις και συστάσεις. Θέλω να γίνει κάποια διόρθωση πορείας κάποιες λύσεις να εξευρεθούν στα πλαίσια των ισχυουσών συνθήκων. Φυσικά και δεν προτείνω κάποια τροποποίηση των συνθήκων. Και έχω προτείνει τα εξή στο κείμενό μου. για την λειτουργία των πόλεων και την εκπροσώπησή τους στα, στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε το θέμα των πόλεων, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει σε σχέση με τη συμφωνία του Άμστερνταμ. Και αναγνωρίζουμε ότι εδώ υπάρχει ένα κοινωτικό κεκτημένο. Οπότε και προτείνουμε οι πόλεις να έχουν πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών. Επίσης, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την εκπροσώπηση των πόλεων στην Επιτροπή των Περιφερειών. Πρώτα-πρώτα έχουμε τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τις πόλεις. Και θα πρέπει να πλησιάσουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτές οι ενώσεις πόλεων, το EuroCities δηλαδή, και οι συναφείς οργανώσεις να είναι κάτι σαν μόνιμος σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και επίσης προτείνουμε να διερευνηθεί το πώς να έχει κάποια όργανα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που να έχει σχέση με τις, έχουν σχέση με τις πόλεις. Να έχει κάποιες μόνιμες ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο και μέσω αυτών να μπορεί να συμβάλλει σε αυτές τις μόνιμες ομάδες εργασίας η πόλη μπορεί να συμβάλλει στη χαράξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Να, πώς θα τις εντάξουμε στο θεσμικό πλαίσιο της πόλης. Τώρα θέλω να δούμε ένα άλλο στοιχείο. Θα δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε αυτές τις μεγάλες δυνατότητες των Πώς αλλιώς. Και πρόκειται για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καινοτόμο. Προτείνω κάτι καινούριο. Έχουν σημαντικές δυνατότητες οι πόλεις. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο βήμα διαλόγου. Στις πόλεις όπου είναι δυνατόν να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάτι τέτοιο. Και μιλώ για τις πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, που έχουν μη κυβερνικές οργανώσεις, εμπειρογνώμονες, εκεί που ήδη υπάρχει κάποια ζήμωση, κάποιος σχετικός διάλογος. Άρα, σε αυτούς τους χώρους, σε αυτά τα φόρα, μπορούμε να αναλύσουμε, μπορούμε να χαράξουμε ευρωπαϊκές πολιτικές. Οπότε έτσι θα εμπλακούν με ακόμη έναν τρόπο οι πόλεις στην ευρωπαϊκή πολιτική. Να δούμε πώς το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει, πώς το Κοινοβούλιο θα ενθαρρύνει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Και αυτό που το κάνουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ήδη έχουν αναλυφθεί από την Επιτροπή των Περιφερειών τέτοιε πρωτοβουλίε μέσω των πρωτοβουλίων των πολιτών. Άρα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε κάποιες, βίλες, σε κάποιες πόλεις συγγνώμη, που να μην είναι αναγκαστικά και πρωτεύουσε. Και έτσι αυτές οι πόλεις να μας δώσουν περισσότερες δυνατότητες για τέτοιο ζήμωση στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνω να ξεκινήσουν 54 τέτοιες πρωτοβουλίες. Δύο φόρα συζήτηση σαν κράτος μέλος. Ποιες είναι και οι πρωτεύουσες αυτές οι πόλεις. Επίσης, τα Δημοτικά Συμβούλια να εμπλακούν γιατί μπορούν να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε αυτούς τους ε, χώρους συζήτησης. Γιατί ε, τα Δημοτικά Συμβούλια είναι κοντά στους ε, πολίτες, στα πανεπιστήμια, στις ενώσεις πολιτών κλπ. Είναι παράγον πλουραλισμού για τις πόλεις τα Δημοτικά Συμβούλια. Οπότε προσπαθούμε το κείμενο με τις προτάσεις που σας είπα. Προσπαθώ να καλύψω αυτή τη διαδικασία της αναβάθμισης του ρόλου των πόλεων για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που παρέχονται από τις πόλεις. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να υπάρξει τέτοια κατανομή των ε, αρμοδιοτήτων. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αυτή η προσπάθεια αφαιρεί αρμοδιότητες από περιφέρειες ή από κράτη. Απλώς αποτελεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή τους. Και έτσι μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του πολιτικού γίνεσθε η πόλη στην Ένωση. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριο Γιασδόφσκι. Ναι, έχουμε σκιώδη ηγητέ. Ή μάλλον έχουμε κάποιου και από οπότε θα πρέπει μια πιέζει ο χρόνο να είστε α, σύντομοι, γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Όλμπριχτ. Κύριε Περέντα, έχετε πρώτα στο λόγο. Ευχαριστώ και πρώτα-πρώτα και τον κύριο Ζεσντόφσκι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε για το, το κειμενό του που περιέχει τόσο ενδιαφέρουσε ιδέες και νομίζω πως είναι σημαντικό σε συνέχεια των όσων είπε να δούμε το πώς θα θεσμοθετηθεί αυτή η εκπροσώπηση και η συμβολή των πόλεων πρώτα μέσα από την Επιτροπή των Περιφέρειων. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε και κάποιο είδους εδαφική συμμετοχή. Δηλαδή ε, να έχουμε περισσότερη συμβολή και είναι άτυπη. Ε, αλλά θα είναι πάρα πολύ σημαντική και έτσι αυτό θα κάνει τη διαφορά. Οπότε θα πρέπει και οι δύο αυτές πτυχές να ληφθούν υπόψη και να σας ε, πω στο ίδιο πνεύμα ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο στο συμπέρασμα στο ότι δηλαδή ακόμα δεν εμπλέκονται αρκετά οι πόλεις ε, και ε, αυτό είναι ένα δύνατο σημείο Οπότε θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί. Όχι, δεν λέω να κάνουμε καινούργια θεσμικά όργανα, απλώ να βελτιώσουμε την αρχιτεκτονική που ήδη υπάρχει. Και ε, υπάρχει ετερογένεια στον χαρακτήρα και στο θεματολόγιο εν μέσω των πόλεων. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει με ενιαίο σχήμα, ενιαίο τρόπος και μέθοδος συνεργασίας. Άρα να γίνει κάποιο είδου άτυπη, ευέλικτη συνεργασία και έτσι οι πόλεις να μπορούν να συμμετάσχουν στην παρασκευαστική διαδρομή μπορούν να μας δώσουν πυρογνωμοσύνη και να διαμορφώσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Οπότε θα πρέπει τα θέματα των πόλεων να βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής της ε, Ένωσης και θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση. Είναι σημαντικό αυτό για τις πολιτικές που άμεσα αφορούν τις πόλεις. Μην έχουμε επικαλύψεις, να έχουμε ζήμωση, να έχουμε διαβούλευση. Το Κοινοβούλιο να προωθήσει όλα αυτά και η Επιτροπή των ε, Περιφερειών θα πρέπει να έχει πρωτογνωστικό ρόλο αλλά θα πρέπει και οι πόλεις να αξιοποιήσουν τα δίκτυα συνεργασίας και έτσι να έχουμε μια πολιτική συνοχή δυναμική μετά το 2020. Θα πρέπει όλα αυτά να τα προτείνουμε, να τα ζητήσουμε. Έτσι να πάμε προς νέα πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Εσείς. Μην ξεχνάτε πιέζει ο χρόνος, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι η σκιώδης εισηγήτρια έχει προετοιμάσει ένα γραπτό σημείωμα το οποίο θα σας μεταφέρω. Θα ήθελα επίσης να κάνω και ορισμένες παρατηρήσεις ε, σαν ε, σοσιαλιστική ομάδα για την έκθεση. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον στενάδελφο Πρέντα και νομίζω ότι έτσι και αλλιώς αυτή είναι και η θέση του εισηγητή. Δεν θα πρέπει να προβλέψουμε να κάνουμε κάποιες θεσμικές αλλαγές, γιατί αν προβλεφθούν θεσμικές αλλαγές είναι σαφές ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα έπρεπε να ονομάζεται Περιφερειών και Πόλεων, αλλά επίσημα η ονομασία είναι αυτή. Πάντως η εκπροσώπηση των πόλεων είναι πολύ ισχυρή και εξαρτάται από τις εσωτερικές θεσμικές ρυθμίσεις σε κάθε χώρα που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει λόγος που ορισμένες χώρες εκπροσωπούν εκπροσώπους πόλεων ε, και άλλοι ε, όχι. Ενώ ας πούμε από τη Γερμανία υπάρχουν εκπρόσωποι από περιφέρειες ή από ε, πόλεις περιφέρειες ενώ στην Ιταλία έχουμε εκπροσώπους και των περιφερειών και των πόλεων και είχαμε και των επαρχιών όταν η επαρχία ήταν θεσμικό η μονάδα. Λοιπόν, αυτό το οποίο μένει είναι ότι για να τροποποιηθεί ακριβώς η ρύθμιση της Επιτροπής ε, ε, των Περιφερειών πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Πάντως στο εσωτερικό των συνθήκων είναι δυνατόν να γίνει μια προσπάθεια για μεγαλύτερη εμπλοκή των πόλεων. Σύμφωνα με την άποψή μου λοιπόν υπάρχει πρώτον ε, μια συζήτηση για τις πόλεις, αλλά στα πλαίσια της επόμενης πολιτικής συνοχής θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο χώρο σε αυτό το οποίο εγώ θα ονομάσω εδαφικές ιδιαιτερότητες. Έχουμε σαν παράδειγμα ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο των πόλεων στην διαχείριση των προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης. Έχουμε επίσης και άλλα εδάφη, τις ορεινές περιοχές, τις απότερες περιφέρειες, ε, τις ε, παράκτιες περιφέρειες με ειδικά χαρακτηριστικά επίσης. Θα πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν στην μελλοντική ρύθμιση της πολιτικής συνοχής να ληφθεί υπόψη μέσω των υπηρεσιών και μέσω των συγκεκριμένων πολιτικών όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι σαφές ότι είναι καλή η ιδέα επίσης και για ένα φόρουμ ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των περιφερειών που έχει πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που οργανώνει το φόρουμ των πόλεων, έτσι ώστε να αποφύγουμε επικαλύψεις. Και αυτό το οποίο έχει σημασία πάντως είναι να υπάρχουν κάποιες στιγμές κομβικές για την Ένωση στα πλαίσια των οποίων να συζητάμε για την πολιτική των πόλεων. Νομίζω ότι επ' αυτού θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι γιατί το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ζει στις πόλεις. Και πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία έχουμε και πάρα πολλές από τις ευκαιρίες τις οποίες έχουμε γεννιούνται και δημιουργούνται στις πόλεις. Θα ήμουν κατά και εγώ της ιδέας επίσημων ή ανεπίσημων ρόλων σε επίπεδο συμβουλίου ή ουδήποτε άλλου θεσμικού οργάνου ειδικά για τις πόλεις. Νομίζω ότι ε, και το Συμβούλιο θα πρέπει να ακούει πιο συχνά τις, ε, τους εκπροσώπους των πόλεων των διαφόρων συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως μιλάμε ειδικά για ένα μοντέλο διαβούλευσης και όχι για συμμετοχικά σχήματα. Νομίζω ότι ξεπεράσατε το χρόνο σας αρκετά. Θα ήθελα να μιλήσουν όλοι οι σκιώδεις και ο κύριος Σόλμπριχτ. Έχουμε πέντε λεπτά συνολικά, γι' αυτό παρακαλώ όσο πιο σύντομα μπορείτε. Κυρία Ρουίση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοί μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι τα θέματα τα οποία συζητιώνται και αποφασίζονται σε επίπεδο της Επιτροπής Περιφερειών. Αυτό το οποίο θα ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο συγκεκριμένο σημείο γιατί πράγματι θα πρέπει να αναζητηθούν δυνατότητες βελτίωσης ε, και επιρροής ε, στις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εκπροσώπων των πόλεων αποφεύγοντας φυσικά οι εσδήποτε μορφές επικάλυψης, διευκολύνοντας τον διάλογο τον οποίο θα πρέπει να περάσουμε και επίσης ξεπερνώντας και τα εμπόδια τα οποία έχουμε. Η ιδέα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ είναι μια πάρα πολύ θετική ιδέα την οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε και να την εντάξουμε στον φυσικό της χώρο την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι σαφές ότι και για το σύνολο των πολιτικών συζητήσεων η Επιτροπή των Περιφερειών είναι κεντρικό σημείο, είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρος για την ολοκλήρωση των πολιτικών συζητήσεων. Θα ήθελα όμως να πω ότι θα πρέπει όλα αυτά τα στοιχεία να ενταχθούν στο εσωτερικό των δομών τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, είναι σαφές ότι θα προχωρήσουμε σε στενή συνεργασία με τον εισηγητή. Τον ευχαριστούμε για τις προτάσεις τις οποίες έκανε και ελπίζουμε να υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα μας βρει συμφώνους. Άντισον. Παρακαλώ πολύ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Δεν πίστηκα ότι υπάρχει ανάγκη να επαναδιαρθώσουμε την Επιτροπή, την ε, Επιτροπή των Περιφερειών, ενσωματώνοντας περισσότερες πόλεις. Γιατί πραγματικά δεν είναι ξεκάθαρο το για ποιους λόγους πρέπει να αλλάξει αυτή η δομή. Μπορείτε να με πείσετε. Δεν πίστηκα ακόμα. Βεβαίως, Προσπαθούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των περιφερειών και των πόλεων. Ίσως πρέπει να ακούσουμε περισσότερο τις πόλεις. Ενώ ήδη οι πόλεις είναι αυτές που εισακούγονται περισσότερο, αυτός είναι ο τρόπος, δεν είμαι πεπισμένος ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Η ευρωπαϊκές πόλεις. Τα δύο φόρουμα ανά χώρα, η εκπροσώπηση πάνω από ένα εκατομμύριο πολιτών μέσω αυτών των πόλεων. Δεν ξέρω ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να υλοποιηθούν αυτέ οι ιδέε. Παραδείγματο χάρη για χώρε όπω η Μάλτα, η Σλοβενία, το Λουξεμβούργο. Δεν είναι σαφέ για μένα τι προτείνεται εδώ. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία των ε, λεπτομεριών. Κύριε Σόλ, είστε σκιώδης. Ναι. Δεν είστε όμως στον κατάλογό μου. Σύντομος παρακαλώ. Ένα λεπτό μας μένει και θέλω να δώσω το λόγο και στον εισηγητή πάλι. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Δύο είναι τα θέματα που θέλω να συζητηθούν. Τι είναι η σχέση μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κοινοτικό επίπεδο και αν θέλετε η, το ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί χρειάζεται περισσότερη επιχειρημασία. Δεύτερον, συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο Άντερσεν. Βεβαίως οι σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών που εκπροσωπούνται περισσότερο οι χώρες και περισσότερο οι περιφέρειες το θέμα της δημοκρατικής εκπροσώπησης, της εκπροσώπησης των πολιτών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Ποιο είναι το καλύτερο επίπεδο, επίπεδο κοινοτήτων και πόλεων, περιφερειών, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Μιλήσατε επίσης και για το φόρουμ και την συμμετοχή, την δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών μέσω αυτών των φόρουμ. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να επεξεργαστούμε πολύ περισσότερο αυτή την πρόταση γιατί είναι ενδιαφέρουσα. Thank Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σύντομο. Κύριε Όλμπριχτ, περιμένετε με υπομονή τόση ώρα. Θα σας ακούσουμε λοιπόν και εμείς με υπομονή. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Την ε, Επιτροπή Ρέτζι, στην οποία ανήκω. Γιατί η ΑΦΚΟ ε, είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Είναι θέμα αύκο αυτό, είναι θέμα αρμοδιότητά σας ή όχι. Ναι, είναι σημαντικό γιατί πρόκειται για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Πρόκειται για κάτι που δεν αφορά τη χρηματοδότηση των πόλεων. Θέλετε να υπάρχει πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Αυτό είναι το ερώτημα. Σαφώς και οι πολίτες απαντούν ναι και η διοίκηση διαφορετικά. Και κυρίως στην Ήπεθρο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τους πολίτες. Η Ήπεθρος και οι περιοχές εκτός των αστικών περιοχών σαφώς και ε, αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικές καταστάσεις στην Ευρώπη. Και βεβαίως εδώ δεν μιλάμε για το θέμα παραδείγματο χάρη του δικτύου των ε, δημάρχων, το οποίο είναι κάτι που το έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι η Επιτροπή των ε, Περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή, παραδείγματο χάρη, που οργανώνει όλε τι πρωτοβουλίε που αφορούν τον πολιτισμό, τι πολιτιστικέ πρωτεύουσε. Πρωτοβουλίε λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τη Επιτροπή των Περιφερειών. Συμφωνώ λοιπόν ότι είναι θέμα που αφορά τη συνθήκη. Η εκπροσώπηση λοιπόν στην Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα θέμα που σίγουρα μπορεί να σας αφορά, αλλά η ισορροπία μεταξύ του τοπικού, του περιφερειακού και εδώ κάνω μια πολιτική πρόταση αν θέλετε, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα που προβλέπεται από τις συνθήκες να αλλάξει αυτή η ισορροπία. Αν αλλάξουν όμως οι συνθήκες, αν αλλάξουν οι όροι και οι προϋποθέσεις, εκεί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι κάτι που αφορά όχι μόνο την Ήπεθρο, όχι μόνο τις περιφέρειες εκτός αστικών περιοχών, αλλά και τις πόλεις. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, λέει ο Πρόεδρος, Σχέδιο θα υποβληθεί το Φεβρουάριο, έτσι λέω. Προθεσμία για τις τροπολογίες. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, διαβάζω το χρονοδιάγραμμα των, ε, της Επιτροπής Ρέτζι. Η προθεσμίες για την υποβολή των τροπολογιών είναι 20 Μαρτίου του 2018. 25 Απριλίου θα επεξεργαστούμε τα, τις ε, τροπολογίες. Αυτές τις προθεσμίες έχω. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει κάτι στα διάφορα. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έδωσα πάλι το λόγο στον εισηγητή, αλλά καταλαβαίνετε γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος της συνεδρίασης. Α, συγγνώμη. 21 Μαρτίου στις 9 το πρωί και στις 3 θα γίνει η επόμενη συνεδρίασή μας.